Ωραία, περνάμε και ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της 104 τροπολογίας. 104. 104 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία τώρα 164. Υπέρ της 164 κατά αποχές εγκρίθηκε. 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 169 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην τροπολογία 177 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στη συνέχεια στην 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 187 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 200... συμβασμός 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 216. 216 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 217 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 218 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 220 υπέρ. Ε, να ελέγξουμε, εντάξει, ελέγχουμε τη 200 18. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 26 εναντίον ε, εγκρίθηκε. 220 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίθηκε. 219 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 226 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 228 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Το ξέρα ναι. 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 238 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 239 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβασμός 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 246 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 247 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 248 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 249 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 250 υπέρ. Τι λέτε εσείς. 249 υπέρ. Ωραία. Και πάλι, τι είπα εγώ, απορρίφθηκε, είπα εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. 249, ωραία. Πέρας ψηφοφορίας λοιπόν τώρα. Καλύτερα είναι να έχει κανεί και μια δεύτερη ματιά. 250 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 251 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 251. Ε, ε, τότε απορρίφθηκε, απορρίφθηκε, τελείωσε. 252 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 253 και 254 ταυτόσημες υπέρ αυτών, κατά, αποχές, απορρίφθηκαν. 255 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 256 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 257 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 258 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. 259 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 260-61 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν. 262 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 263 υπέρ κατά αποχές Απορρίφθηκε, μάλιστα. 265 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίθηκε. 266 υπέρ. Με προφορική τροποποίηση. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 267 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 270 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 273 υπέρ. Κατά τι λέτε εσείς. Ε, τότε να ακούτε την ε, πολωνική μετάφραση. Πάρετε την πολωνική μετάφραση. Ε, βασίζεσαι στο, στη γερμανική μετάφραση. Δεν ε, εμπιστεύεστε την Ίζα. Τι γίνεται. 273 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 274 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 276 υπέρ. Όχι, καλύφθηκε λέει αυτή. 276 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 282 υπέρ, εγκρίθηκε. 281 Εντάξει, τη 277 τώρα λέγεται στον πρόεδρο. 77 και 282, επιλέξτε ποια θέλετε. Ολοκληρώθηκε. Εντάξει. Πάει. «281. Ο κύριος Τάνοκ επέλεξε τη λάθος τοπολογία. 281. Ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 283. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Μου φαίνεται ότι εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 291. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 32 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε και άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά επί της 32. 32, έτσι. Πέρας ψηφοφορίας λοιπόν τώρα. Μάλιστα. Απορρίφθηκε με ισοψηφία. Απορρίφθηκε. Περνάμε στο συμβασμό 6 υπέρ. Κατά Χέσα εγκρίθηκε. Και τώρα πάμε στη 42 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 44 όχι 45 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 59 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 60 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 61 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 62 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 8 μια στιγμή, Πρόεδρε, μια στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποβάλω, να προτείνω μια προφορική τροποποίηση. Διαβουλεύτηκα με τους σκιώδεις εισηγητές και προτείνεται, προτείνουν <clears throat> ως υποσημείωση στον συμβιβασμό 8 να αναφέρουμε πολιτικούς κρατούμενους στην Λευκορωσία. Μιχαήλ Αουτοκόβιτς, Μιχαήλ Στετκέβιτς, Ντασκέβιτς, Εντουάρτ Λόμπαου, Άλες Dziadok, Alinevich, Αλεξάνδρ Φρανσκέβιτς. Αυτά είναι τα ονόματα των πολιτικών κρατουμένων στην Πέλαρους που θέλουν να αναφέρονται στην υποσημείωση. Ως υποσημείωση λοιπόν, εντάξει. And the list of political και ο κατάλογος πολιτικών κρατουμένων συμπεριλαμβάνει τα ονόματα αυτά, τα οποία μόλις σας διάβασα, εντάξει. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Με αυτή την υποσημείωση, ποιοι είναι υπέρ του συμβιβασμού 8. Κατά, αποχές εγκρίθηκε. Εντάξει, ποια είναι η τροπολογία επόμενη. Επόμενη τροπολογία 74, μάλιστα. 74. Ποιοι είναι υπέρ της 74, κατά αποχές εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε η τροπολογία 4, τι έγινε με αυτήν. Ωραία, πάμε στην 76, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 77 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 80 υπέρ κατά αποχές και πάλι 80 και πάλι 80 υπέρ κατά αποχές κατά λέει ο πρόεδρος τώρα με αυτόν τον τρόπο διασφάλισα ότι η πλειοψηφία ήταν υπέρ εγκρίθηκε εγκρίθηκε 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τι έγινε με την 81, εγκρίθηκε αυτή έτσι. Πάμε στην 90 τώρα, τροπολογία 90 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 94 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τώρα citations 1 αιτιολογική σκέψη 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και αυτή. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της σύστασης όπως τροποποιήθηκε. Πέρας ψηφοφορία τώρα. Συγχαρητήρια λοιπόν, συγχαρητήρια κύριε Παλέσκης για την έγκριση της πρότασης ε, σύστασης. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο είναι η ενημέρωση από τον Πατεκό Γκάλαχερ για την έκτη συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισλανδίας που έλαβε χώρα στο Ρέικεβικ της Ισλανδίας και πρόταση ψηφίσματος για την έκθεση πρόοδου 2010 για την Ισλανδία και τις προοπτικές μετά τις εκλογές. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 4η Σεπτεμβρίου 2013 στις 12 το μεσημέρι. Δίνω το λόγο αμέσως στον κύριο Πατεκόπ Γκαλαχέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απευθύνω την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα τη συνάντησή μα στην Ισλανδία την περασμένη εβδομάδα. Όπω θα γνωρίζετε όλοι, οι βουλευτικέ εκλογέ έλαβαν χώρα στην Ισλανδία στι 27 Απριλίου και σήμερα έχει εγκαθιδρυθεί μια νέα κυβέρνηση στην Ισλανδία, η οποία πάγωσε τι ε, διαπραγματεύσει ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δήλωσε ότι η συνέχιση θα εξαρτηθεί από δημοψήφισμα. Υπάρχει λοιπόν μια αλλαγή πολιτικής κατάστασης στην Ισλανδία η συνείδηση της κοινή κοινοβουλευτική Επιτροπής στις 27 Ιουνίου στο Ρέικιαβικ μεταξύ Ισλανδία και Ευρωπαϊκή Ένωση. έλαβε χώρα με επίσκεψη σε δύο χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα και συναντήθηκαμε και με διάφορου Οργανισμού. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε καλύτερα τη νέα προσέγγιση της Ισλανδικής κυβέρνησης όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσει προσχώρηση και προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα των απόψεων των διαφόρων πολιτικών κομμάτων καθώ και διαφόρων τμήματων τη κοινωνία. Να σα συνοψίσω τι διαπιστώσει μα. Τα κόμματα του συνασπισμού, ε, το φιλελεύθερο και οι προοδευτικοί επικύρωσαν την στάση τους κατά της πρόσβασης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης παραμένουν χωρισμένα, αλλά φαίνεται να είναι υπέρ της ολοκλήρωσης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Υπάρχει αυτή η όλο και λιγότερη διάθεση προσχώρησης λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και οι διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισλανδίας για διάφορα θέματα. Αφού λοιπόν τέθηκαν σε αναστολή οι διαπραγματεύσεις, θα προχωρήσουμε σε μια αξιολόγηση των διαπραγματεύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα παρουσιαστεί στο Ισλανδικό Κοινοβούλιο, αναμένεται το φθινόπωρο. Παραμένουν εκκρεμή ερωτήματα όσον, αφορά την νέα προσέγγιση της Ισλανδικής κυβέρνησης σε σχέση με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Οι συζητήσεις κατά το JPC ειδικότερα μας επιβεβαίωσαν τις αμφιβολίες που έχει η κυβέρνηση ότι μπορεί να μην γίνεται εν ψήφισμα δημοψήφισμα και αυτό φαίνεται πιθανό ότι αυτή η κυβέρνηση που είναι κατά της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις ακόμη και αν ψηφίσει υπέρ ε, το Κοινοβούλιο. Τώρα το σε ποιο βαθμό θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην υλοποίηση της απόφασης παγώματος των διαπραγματεύσεων δεν είναι σαφές. Δεν είμαστε σίγουροι τι θα συμβεί με την υλοποίηση του ενταξιακού μέσου ή τα έργα IPA. Η νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε μετά τις εκλογές ε, ότι θέλει να ανασταλούν όλα τα προγράμματα. Αλλά αυτό, όπως είπα, παραμένει υποσυζήτηση. Μια τέτοια απόφαση θα οδηγήσει σε οπισθοχώρηση όσον αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Η Ισλανδία, λοιπόν, συνεχίζει να θέλει να διατηρεί στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλους τομείς, να ενισχύσει και να εμβαθύνει τις σχέσεις σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Η νέα κυβέρνηση θεωρεί τον ΕΟΧ ως την κύρια πλατφόρμα για τέτοιου είδους συνεργασία. Ένας άλλος τομέας συνεργασία είναι το ΑΡΤΕΚ που συζητήσαμε επίση στη συνάντηση JPC. Η Ένωση και η Ισλανδία ε, θέλουν να επιταχύνουν τη συνεργασία σε αυτό το τομέα με έναν ε, διάλογο υψηλού επίπεδου για τα θέματα της Αρκτικής. Αυτός ο διάλογος θα ε, συνεχιστεί Όσον αφορά τη διανοίξη μακρό, η Ισλανδική κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν θα βοηθήσουν οι κυρώσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βουλευτές ε, αμφισβητούν την ομιμότητα τυχών κυρώσεων. Φυσικά αυτό θα το μάθουμε μέχρι την υλοποίηση των κυρώσεων. Αυτό συζητήθηκε επίσης και στη συνάντηση με τους ε, οργανισμούς εκπροσώπων και ορισμένοι εκπρόσωποι των Ισλανδών μας έκαναν έκκληση να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο και να διευκολύνουμε τις συζητήσεις για το, για το Μάκρο. Υπήρξαν πολύ δραστήριες συζητήσεις, πολύ ζωντανές για να προδεύσουμε σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ε, λοιπόν, η προσέγγιση αυτή τη νέα κυβέρνηση για τις ενταξιακές διαπραγματεύσει παραμένει αμφισβητήσιμη. Περισσότερε ερωτήσει έχουν μείνει παρά απαντήσει. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και αν θα γίνει δημοψήφισμα. Η υλοποίηση της απόφασης παγώματος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων έχει συνέπειες για την προενταξιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει να αξιολογηθεί σε περισσότερο βάθος. Η νέα προσέγγιση λοιπόν χρειάζεται σαφώς τεχνικές και φυσικά πολιτικές απαντήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς συμφωνήσαμε να κάνουμε τη δεύτερη μα συνάντηση φέτος, 27 και 28 Νοεμβρίου και εγώ αναμένω ότι στο μεταξύ θα έχει δημοσιευτεί η αξιολόγηση της κυβέρνησης για τις διαπραγματεύσεις και τις εξέλιξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά μέλη εδώ ήταν παρόντας, εκείνες τις συναντήσεις ε, και ο Τέιλερ και ο Σπίτσεν Πρέντα και μπορούν να σας επιβεβαιώσουν την τρέχουσα κατάσταση. Ευχαριστώ. Ε, now I pass the floor to... Τώρα δίνω το λόγο στον, στον εισηγητή, κύριο Παρέντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, εάν συμφωνείτε κι εσείς, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την ε, έκτη συνάντηση της ε, κοινή Κοινοβουλευτικής Συνόδου ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισλανδίας. Καταρχάς να σημειώσω ότι η υποδοχή ήταν εξαιρετική στην Ισλανδία. Συναντήσαμε πέντε πολιτικούς αρχηγούς από τους έξι που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Οικονομικών, ε, που είναι και ηγέτες των πιο σημαντικών πολιτικών ε, ομάδων, ε, κομμάτων δηλαδή, που ηγούνται του κυβερνητικού συνασπισμού. Δεν θέλω να πω όμως και κάτι άλλο, το δεν θέλω να το λάβετε σαν κακή παρατήρηση. Στην αρχή η πολιτική, το πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκει ο Πρωθυπουργό ήταν υπέρ της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Πρωθυπουργό μιλάει για την προσχώρηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για το ψήφισμα τώρα, αποφασίσαμε ε, για το ότι το ψήφισμα που θα αφορά την Ισλανδία θα ε, ε, αναβληθεί. Να σας υπενθυμίσω ότι συζητήθηκε το θέμα στο, στην Ολομέλεια και ήταν, είχε διαμορφωθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Δεν μπορούμε απλώς και μόνο να ε, αναφερθούμε στο τι έγινε για το 2012 λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις, ε, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Οι διαπραγματεύσεις ε, έχουν σταματήσει. Γι' αυτό ακριβώς ελήφθησαν δύο αποφάσεις. Το ένα είναι να τροποποιήσουμε το ψήφισμα καταρχήν και δεύτερο να έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο κείμενο το οποίο να συνοψίζει την νέα πολιτική κατάσταση, την πολιτική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί δηλαδή μετά τις ε, εκλογές. Η πρώτη απόφαση είναι να προσθέσουμε στον τίτλο, εκεί που λέγεται την πρόοδο για το 2012, στον τίτλο να αναφέρουμε και τις μετεκλογικές προοπτικές στην Ισλανδία. Διαναλάβουμε υπόψη μας δηλαδή και τις συνθήκες που μας ανάγκασαν να αλλάξουμε την, ε, τους όρους της συζήτησης. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το μετεκλογικό, μετεκλογικές προοπτικές θα πρέπει να ε, αναφερθούν, να αναφέρεται στον τίτλο, διότι και στο κυβερνητικό συνασπισμό ούτως ή άλλως υπάρχουν δύο κόμματα τα οποία είναι κάθετα αντίθετα στην ε, προσχώρηση της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση τονίσαμε αυτό το θέμα, ο, τονίστηκε αυτό το θέμα, δηλαδή ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν θέλει να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις ε, εάν και εφόσον δεν οργανωθεί πριν ένα δημοψήφισμα. Και το δημοψήφισμα θα πρέπει να έχει το εξής ερώτημα. Θα πρέπει ή να συνεχίσουμε ή όχι τις διαβουλεύσεις. Όμως Ακόμα δεν έχει καθοριστεί ούτε η ημερομηνία του δημοψηφίσματος, ούτε το περιεχόμενό του ακριβώς. Γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν βιάζεται ιδιαίτερα να προχωρήσει, γιατί από ό,τι φαίνεται θέλει πρώτα να γίνει μια ζήτηση στο Κοινοβούλιο, το φθινόπωρο, και να γίνει μια αξιολόγηση της κατάστασης και όπως προχωρούν διαβουλεύσεις και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ρέκεβικ μας είπαν ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ενδεχόμενα να γίνει αυτή η συζήτηση και μετά τη συζητήση στο Κοινοβούλιο θα υπάρχει ενδεχόμενα η δυνατότητα να ληφθεί μια απόφαση που θα είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνει το δημοψήφισμα το 82% του πληθυσμού φαίνεται ότι θέλει το δημοψήφισμα αυτό να οργανωθεί ταυτόχρονα με τις τοπικές εκλογές που θα λάβουν χώρα το 2014. Επομένως φαίνεται ότι μπορεί μεν το δημοψήφισμα να είναι ένα θέμα αμφιλεγόμενο στην Ισλανδία, οι περισσότεροι Ισλανδοί όμως θέλουν να γίνει ένα τέτοιο δημοψήφισμα που θα αφορά τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Τώρα, από ό,τι φαίνεται οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία, το 60% περίπου των ε, Ισλανδών θέλουν να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Το 40% θέλει να σταματώσει. Επομένως στο ψήφισμα ε, θα συμπεριλάβουμε ε, συμπεριλαμβάνουμε μάλλον την πρόταση που λέει ότι θα έπρεπε η Ισλανδική κυβέρνηση να περιμένει το πέρα στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και μετά να οργανωθεί το δημοψήφισμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρετε, είχε υποδεχθεί με ενθουσιασμό το αίτημα προσχώρησης ε, της Ισλανδίας. Και ο Πρωθυπουργός ε, είχε ε, εκφράσει τη δέσμευσή του για να προχωρήσουν τα πράγματα. Είχαν ξεκινήσει, είχαν ανοίξει 23 κεφάλαια ήδη και θα ήθελα να ζητήσω, να ρωτήσω από τους συναδέλφους να κάνουν κάποιες προτάσεις, προτάσεις βελτίωσης της έκθεσης εγώ πιστεύω πάντως ότι το κείμενο το δικό μας πρέπει να είναι συγκεκριμένο και θα πρέπει με ένα συγκεκριμένο και ε, τρόπο να ε, αναφέρουμε τους στόχους μας δεν νομίζω ότι μπορούμε να κεντήσουμε εδώ από αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μεγάλο, ένα μεγάλο κείμενο. Και στο κάτω-κάτω υπάρχει και η έκθεση τη ε, προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις ήταν ε, ε, καλέ, αλλά τελείωσαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Φάμ, ποια είναι η άποψή σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Πρέντα για το πολύ ισορροπημένο κείμενο του μετά την αλλαγή κυβέρνηση στην Ισλανδία η δουλειά του πρέπει να ήταν πολύ δύσκολη. Το κατανοώ. Ευχαριστούμε επίση και την Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα σχόλιά του περί της κατάστασης, επειδή πραγματικά τώρα πρέπει να αξιολογήσουμε την τρέχουσα κατάσταση. Το να έχουμε μια υποψήφια χώρα που παγώνει τι ενταξιακέ διαπραγματεύσει, είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο. Πιστεύω πρέπει οπωσδήποτε, ανεξάρτητα από το πόσο δεν μα αρέσει η θέση τη νέα κυβέρνηση. είμαστε υποχρεωμένοι να τη σεβαστούμε και να μην του εξασκήσουμε υπερβολική πίεση. Οι δράσεις της Ισλανδικής κυβέρνησης είναι λυπηρές. Πολλοί και από την ομάδα μου και άλλοι θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι να υποδεχθούμε μια τέτοια χώρα με έντονη δημοκρατία και ισχυρού θεσμού και ε, κατά βάση ισχυρή οικονομία. Ωστόσο, η Ισλανδική κυβέρνηση είναι εκείνη που θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα και εμεί είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε την άποψη του Ισλανδικού λαού. Ωστόσο, πρέπει να αξιολογήσουμε αυτή την κατάσταση και να βρούμε έναν επικοδομητικό ισορροπημένο τρόπο για να συνεχίσουμε. Η Ένωση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κλείσει τις πόρτες. Πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτό το φάκελο της αίτησης μέλους της Ισλανδίας και να μην οθήσουμε ή πιέσουμε την Ισλανδία ώστε να μας δώσει ένα οριστικό ναι ή όχι. Ας μην προκαλέσουμε μια αρνητική αντίδραση εξασκώντας υπερβολική πίεση. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποδειχθεί ανταπαραγωγικό και να οδηγήσει σε τερματισμό μόνιμο της ε, ενταξιακής διαδικασίας. Ας μην το πράξουμε αυτό. Εκτιμώ ιδιαίτερα την έκθεσή σας, ωστόσο πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε τις παραγράφους 6 και 7, να μην θεωρούμε ότι το δημοψήφισμα είναι δεδομένο και να μην πιέσουμε γι' αυτό. Οι συζητήσει στην Ισλανδία σήμερα δείχνουν ότι εφόσον δεν έχει οριστεί η ημερομηνία, εξακολουθεί να υπάρχει το ενδεχόμενο άλλων επιλογών από ένα γρήγορο δημοψήφισμα. Σίγουρα αμφισβητούν ε, το πόσο επωφελές θα είναι οι δύο μέλους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να μην θέλουν να προχωρήσουν αυτή τη στιγμή, αλλά αν η κυβέρνηση είναι της άποψης ότι ένα προσωρινό πάγωμα της ενταξιακής διαπραγμάτευσης μπορεί να γίνει χωρί χωρίς δημοψήφισμα, ίσως αυτή είναι μια καλύτερη επιλογή, επειδή όπως είπε και ο κύριος Γκάλαχερ, κάτι πιο οριστικό θα δημιουργήσει διάφορα προβλήματα για τα διάφορα τρέχοντα προγράμματα, για τις συζητήσεις, για τις διάφορες διανέξεις, για όλα αυτά τα θέματα, τίποτα καλό δεν θα μπορούσε να προκύψει από ένα άμεσο δημοψήφισμα. Ας παραμείνουμε λοιπόν σε στενή επαφή με τους Ισλανδούς, ας κρατήσουμε ανοιχτό το διάλογο για εμάς το να γίνουν μέλη ε, είναι ένα πολύ σημαντικό ε, θέμα που μας αφορά ιδιαίτερα να τους κρατήσουμε λοιπόν κοντά μας. Ευχαριστούμε κύριε Φαν... Να... Η προθεσμία δεν έχω κανένα άλλο στο κατάλογό μου να σας υπενθυμίσω πότε είναι η ημερομηνία για την υποβολή των τροπολογιών. Α, όχι. Κάποιον ε, έχασα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήμουνα ένα από τα ευτυχή μέλη της αντιπροσωπείας και είχα την ευκαιρία να προεδρεύσω την Παρασκευή την συνάντηση με τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών στην συνάντηση εκείνη η, η εντύπωση των πολιτών, η εντύπωση που πήραμε από τους πολίτες ήταν ότι θέλανε να συνεχίσουν οι διαβουλεύσεις και συμφωνεί με τον προηγούμενο, συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή ότι θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε τα θέματα αυτά πάρα πολύ προσεκτικά Ε, θα πρέπει να περιμένουμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη ε, συνεργασία ανάμεσα στα δύο βασικά κόμματα. Η συζήτηση που θα λάβει η χώρα στο Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο είναι πάρα πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι τα πράγματα είναι ακόμα ανοιχτά και η συνάντηση της 26-27 Νοεμβρίου θα είναι πάρα πολύ σημαντική από ό,τι είπαν και οι Ισλανδοί συνάδελφοι θα έχουν τότε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Θα ήθελα να σημειώσω και το εξαιρετικό έργο των υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων ε, εκεί. Ε, γιατί οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες ε, και θα πρέπει να αποτίσουμε να φόρο τιμής στην, στη συνεργασία τους. Επισκεφθήκαμε αρκετά project ε, όχι, εγώ δεν μπόρεσα ε, να τα δω όλα γιατί έπρεπε να πάρω το αεροπλάνο μου, ε, το αεροπλάνο μου αλλά πιστεύω και από τους συναδέλφους ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω. Κύριε, ο κύριος Πλέντε να απαντήσει. Δεν είναι μια απάντηση, απλώς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της σοσιαλιστικής ομάδας που κάνανε παρατηρήσεις ε, πάρα πολύ ε, χρήσιμες, για το διάλογο. Θα ήθελα να προσθέσω μια παρατήρηση, μια παρατήρηση που έχει ένα πιο πολιτικό χαρακτήρα, αν μου επιτρέπετε, διότι το ερώτημα, του, το θέμα του δημοψηφίσματος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, κυρίως γιατί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είπε ότι δεν κάνουμε ένα περαιτέρω βήμα στις διαπραγματεύσεις χωρίς το δημοψήφισμα. Αυτό είναι το, ε, το πρώτο που ελέγχθη. μετά όμως ταυτόχρονα είδαμε ότι η κυβέρνηση, η κυβέρνηση είδε ότι οι πολίτες θέλουν ε, να προχωρήσουν στην προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα βρίσκεται, αν θέλετε, η κυβέρνηση παγιδευμένη, διότι ε, Εάν κάνουν το, το δημοψήφισμα υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο πληθυσμό οι πολίτες να πούνε ναι, ε, ενώ η κυβέρνηση είναι κατά της προσχώρηση. Επομένω, ε, από πολιτική πλευρά ε, εδώ τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα του Κοινοβουλίου, του Κοινοβουλίου της Ισλανδίας. Η κυβέρνηση θα επανακαθορίσει τη θέση της και θα ζητήσει από το Κοινοβούλιο να κάνει ακριβώς το αντίθετο αυτό που έκανε στην αρχή, δηλαδή να ξεχάσουμε λίγο τις, να ξεχάσουν τις δια, ε, διαπραγματεύσεις. Είναι πολιτικό το θέμα βέβαια το, με, τις, τα πολιτικά κόμματα της Ισλανδίας. Οι σοσιαλιστές είναι ενθουσιασμένοι με την προσχώρηση. Ε, τα άλλα κόμματα εδιστάζουν κάπως. Πάντως είναι περίπλοκο το θέμα, επαναλαμβάνω, γι' αυτό συμφωνώ με τους σοσιαλιστές συναδέλφους όταν λένε ότι θα πρέπει να ε, προσέξουμε και τις ε, αντιδράσεις στο κείμενό μας. Γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί να, το, να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Επόμενο σημείο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό του 2014, όλα τα τμήματα, η εισηγητής Χωσέ Ιγνάσιος Αλαφράνκα Σαντσονέιρα. Έχετε το λόγο. Sí, gracias, señor Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα θυμόσαστε ότι στην πολιτική συμφωνία που ψήφισε στην Ολομέλεια του Στρασβούργου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικυρώσαμε αφού ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα μας από τα αιτήματα που έχουμε υποβάλει στο Συμβούλιο των Υπουργών που εκφράστηκαν στο πολιτικό ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, θέλω να υπενθυμίσω επ' αυτού ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χρηματοοικονομικό πολιετές πλαίσιο, η αύξηση που προβλέπεται για την εξωτερική πολιτική στο σύνολό της, στο σύνολο των δράσεων των ετών των δημοσιονομικών αυτών προοπτικών, ήταν 3% συνολικά. Αύξηση σε διαφορά με άλλες δραστηριότητες της Ένωσης που περικόπηκαν στα κονδύλια για αυτές αύξηση 3%. Κατά το έτος 2014 που είναι η πρώτη χρονιά των νέων δημοσιονομικών προοπτικών και αξιοπερίεργο είναι ότι η Επιτροπή υποβάλλει μια μείωση πολύ αξιοπρόσεκτη των κονδυλίων για την εξωτερική πολιτική του 12,5%. Για να υπάρχει λοιπόν μια ιδέα από πλευρά για το τι συμβαίνει, ο υπολογισμός σε σχέση με τα κονδύλια δεσμεύσεων υποχρεώσεων το 2013 ήταν ε, ε, ένα συγκεκριμένο ποσό. Το ποσό που προτείνει τώρα για το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 8 δισεκατομμύρια 150 εκατομμύρια. Όπως σας είπα έχουμε μία μείωση 12,5%. Ε, ε, θα κατανοήσετε αγαπητοί συνάδελφοι ως ε, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ότι εγώ ως αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής δεν μπορώ με κανένα τρόπο να συμφωνήσω με μια τόσο σημαντική περικοπή σαν αυτή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αληθεύει τώρα ότι η αύξηση του 3% καθ' όλη την περίοδο, πολυετή περίοδο είναι δεδομένη, αλλά δεν θα είμαστε στο ύψος ε, σε σχέση με τα όσα θέλουμε να χρηματοδοτηθούν ούτε στο ύψος των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πεδίο των εξωτερικών δράσεων αν δεχθούμε αυτές τις περικοπές που είναι τόσο σημαντικές σαν αυτές που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού. Εσείς ακούσατε σήμερα το πρωί τον Υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας που μας έκανε λόγο για την προτεραιότητα που δίνεται στη Σύνοδο Κορυφής της Βίλνιους και όλα όσα αναφέρονται στην πολιτική γειτονία σε σχέση με τις χώρες του Βορρά και τις χώρες της Ανατολής. Και θα ακούσατε και σε σχέση με την Αραβική Άνοιξη που μας ανέφεραν για την κατάσταση στην Αίγυπτο, στη Συρία και σε άλλες χώρες που πλήττονται από αυτή την κατάσταση ε, αστάθειας. Πώς μπορούμε να δεχθούμε τούτων όλων ε, αναφερόμενων μια τέτοια περικοπή για την πολιτική γειτονία του 17% για την πολιτική προένταξης. Κάνουμε λόγο αυτή τη στιγμή για την ε, περίπτωση της Ισλανδίας περίπτωση μείωσης 3,5% του μέσου σταθερότητας και 20,70% για τις δράσεις στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Γι' αυτό η δική μου πρόθεση πρόεδρε είναι και κατανοώ ότι είναι μια τακτικής υφής τοποθέτηση να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε αυτά τα κονδύλια να ενταχθούν στο επίπεδο του έτους 2013 και έχουμε και κάποιες δυσκολίες διαδικαστικές. Αυτές οι διαδικαστικές δυσκολίες έγκυνται στο ότι λόγω των περιορισμών που υπάρχουν που μας επιβάλλονται από την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει να καλύψουμε την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών προτού τοποθετηθεί το Συμβούλιο εφόλων αυτών. Δυστυχώς μίλησα απόψε με την Γενική Συγήτρια του Ευρωκοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό 2014. Εξέφρασα τη δική μας δυσαρέσκεια για τον γεγονός ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με αυτή τη βάση, αλλά μου διασφάλισε ότι θα προσπαθήσει στο μέτρο του εφικτού και είναι πολύ περίπλοκες οι διαπραγματεύσεις, θα προσπαθήσει να ληφθούν υπόψη οι τοποθετήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, οι επιθυμίες αυτής της Επιτροπής. Λίγη στις 16 Ιουλίου η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Ελπίζω να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου τελεσίδικα επ' αυτών. Και αν πρέπει να προσαρμόσουμε τα πράγματα σε σχέση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου των Υπουργών, ελπίζω ότι θα μπορέσει να γίνει με κατάθεση ε, τροπολογιών. Έχω την πρόθεση, Πρόεδρε, προτού ξεκινήσουν οι διακοπές για το καλοκαίρι, αύριο, αν είναι δυνατόν, να συγκαλέσω μια συνάντηση σκιωδών εισηγητών για να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε με αυτή τη στρατηγική και να δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε και για τα κονδύλια. Και η κυρία Γιάτεν που είναι παρούσα και είναι είναι σκιώδης εισηγήτρια της ε, φιλελεύθερης ομάδας. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε Πρόεδρε. Ως μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να δεχθούμε αυτές τις σημαντικές περικοπές είναι απαράδεκτο για την πολιτική εξωτερικών δράσεων που αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο σαν μια πολιτική που έχει αύξηση δραστηριοτήτων δεν μπορεί να αποτελεί μέρος αυτών που εμείς επιθυμούμε κάτι τέτοιο. Και ως προς αυτό είμαι στη διάθεση των συναδέλφων φυσικά για να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τα μελήματά τους τις επιθυμίες τους και να δημιουργηθεί το δημοσιονομικό πλαίσιο με τέτοιο τρόπο παρότι είναι περιορισμένο λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλαφράνκα. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Κανείς δεν ζητάει το λόγο. Επομένως, θα σας είπε... Α, όχι, κυρία Γιατεμάκια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ εξοικονομούμε και τον χρόνο ομιλία μας από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, καταρχάς να πω ότι συμφωνώ με το γεγονός ότι η Κομισιό θέλει να αντιμετωπίσει με έναν ορθολογικό τρόπο τις δεσμεύσεις, διότι στο παρελθόν η Κομισιό αυτή την περίοδο, σε αυτή την περίοδο του έτους υποσχόταν πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούσε να ε, υλοποιήσει τις υποσχέσεις. Θα πρέπει και για τις δεσμεύσεις ε, η δημοσιονομική διαδικασία να ξεκινά πάρα πολύ προσεκτικά, διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι προοπτικές περιορίζονται κατά 12,5% και θα ήθελα να ρωτήσω και την Κομισιό τους εκπροσώπους της Κομισιόν, τι θα γίνει με την ε, πολιτική γειτονίας προς τις ανατολικές χώρες, διότι εκεί οι περικοπές είναι ακόμη πιο δραστικές. Ανέρχονται περίπου στο επίπεδο του 30%, ενώ σε, προς τον Νότο εκεί έχουμε αύξηση ε, των ε, πόρων, των κονδυλίων λίγο βέβαια, αλλά παρόλα αυτά έχουμε ε, αύξηση. Τώρα, για τις ε, αναλήψεις υποχρεώσεων θα πρέπει να ακούσουμε κάποιες ε, εξηγήσεις όσον αφορά τις περικοπές, τουλάχιστον για τις σημαντικές περικοπές επίσης για την πολιτική που αφορά την, τον αρκτικό κύκλο. Τι θα γίνει εκεί, πώς θα χρηματοδοτηθούν ε, οι πολιτικές. Αυτό το κέντρο πληροφοριών της Αρκτικής, πώς θα χρηματοδοτηθεί. Και εν κατακλείδη ήθελα να πω ότι κατανοώ απόλυτα ότι όταν ε, έχουμε περικοπές των πόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε πού θα δοθούν τα χρήματα, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει να τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά, να έχουμε, να, ε, να έχουμε ε, επενδύσεις που θα αποδώσουν, αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα ήθελα να ξέρω και τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, τι αποτέλεσμα είχαν σε, έγιναν σεβαστοί οι στόχοι του Κοινοβουλίου. Η Γκόμες. Κύριε Πρόεδρε, η συγγύτρια κυρία Μαρία Μουνής δεν είναι εδώ, αλλά μου άφησε μερικές σημειώσεις που αποτυπώνουν τις δικές της ανησυχίες και συνεπώς της ομάδας μου. σχετίζονται με το κύριο μας, ε, την κυρία μας ένσταση στην Επιτροπή που αφορά την υποχρηματοδότηση της επικεφαλίδας 4 κάθε χρόνο στον προπολογισμό φέτος όταν οι προβλεπόμενες περικοπές φτάσουν το 10,5% περισσότερο από ότι στον προϋπολογισμό του 2013 πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πάνω απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε, να μας προβληματίσει το γεγονός κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον προπολογισμό μπορεί να γίνει ο παγκόσμιος φορέας επιρροής που θέλουμε να είναι σε αυτή την Επιτροπή. Επίσης θα θέλαμε όλοι οι συναδελφοί να αντιληφθούν ότι αυτή η τεράστια περικοπή είναι συνέπεια του MFF του 2014 μέχρι 2020 που είναι ανεπαρκές και στερείται φιλοδοξίας. Η συμφωνία που επετεύχθη για τις μειώσεις του MFF όπως γνωρίζετε 16% από την αρχική πρόταση της Κομισιόν για ολόκληρο το διάστημα. Εμάς μας ανησυχούν ιδιαίτερα οι προτινόμενες περικοπές για το ENI 14,5% λιγότερο και για το DCI με μείωση του του 12,6% και τα δύο αυτά είναι προτεραιότητες όχι μόνο για τη δική μας ομάδα αλλά πιστεύω, πιστεύουμε για ολόκληρη την Επιτροπή Συμμεριζόμαστε λοιπόν την άποψή του εισηγητού του κ. Σαλαφράγκα και προτείνουμε τροπολογίε ώστε να ενισχύσουμε την αντίθεσή μα σε έναν προπολογισμό που σε πολύ σημαντική μείωση, υποβάθμιση του ρόλου μα. Ε, κύριε Σαλαφράγκα. Κύριε Σαλαφράγκα, ευχαριστώ πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά τις παρατηρήσεις της κυρίας Γιάτεν Μέκη από τις ερωτήσεις που τόσο νόμιμα έθεσε, οι ερωτήσεις στρέφονται ουσιαστικά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ θα ήθελα να συμμεριστώ αυτές τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Να ακούσουμε την Επιτροπή και μετά να απαντήσω και να τοποθετηθώ απαντώντας στις ανησυχίες της συναδέλφου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε συνάδελφε. Υπενθυμίζω η προθεσμία για τις τροπολογίες ε, για την γνωμοδότηση πριν του προπολογισμού 16 Ιουλίου 12 το μεσημέρι να σημειωθεί ότι μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες μόνο στην αγγλική γλώσσα. Και προθεσμία για τις ε, δημοσιονομικές τροπολογίες είναι και πάλι 16 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι αλλά μπορείτε εκεί να υποβάλλετε τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες. Παρακαλώ κύριε Σαλαφράγκα. Πρόεδρε, δεν είναι ότι δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ, είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της Επιτροπής που θα μπορούσε να απαντήσει στις ανησυχίες που εξέφρασε η κυρία Γιάτεν Μέκη και που επιμένω, συμμερίζομαι εγώ προσωπικά. Καλό και ευκταίο θα ήταν να μπορέσουν να μας δώσουν τις ε, απαντήσεις τους ε, μπροστά στις αμφιβολίες που διατυπώθηκαν εδώ. Η Επιτροπή μπορεί να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή εδώ δεν έκανε τίποτα άλλο από το να υλοποιήσει την απόφαση για τα ανώτατα όρια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Η μείωση αυτή του 12,5% των πιστώσεων σε σχέση με το 2013 οφείλεται απλά και μόνο στο γεγονός ότι το ανώτατο όριο του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2014 μας περιορίζει. Σε αυτό το ανώτατο όριο Σα υπενθυμίζω ότι η Κομισιόν το 2011 είχε προτείνει αύξηση τη επικεφαλίδα 4 της τάξη του 20% νομίζω στην πρόταση του 2011. Η πρόταση της Κομισιόν μειώθηκε σχεδόν κατά 20% στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Η εν λόγω μείωση οδηγεί λοιπόν σε μείωση του 12,5% στο 2014 σε σχέση με το 2013. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει μια πρόταση η οποία να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του δημοσιονομικού πλαισίου. Προτείναμε ένα περιθώριο των 152 εκατομμύριων ε, για τις δημοσιονομικές προεπτικές που είναι αρκετά μεγάλο περιθώριο δεδομένα των περιορισμών. Χρειάστηκε λοιπόν να αποτυπωθούν αυτές οι περικοπές του δημοσιονομικού πλαισίου σε σχέση με τις αρκετές προτάσεις για τα κονδύλια σε όλα τα μέσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κοινοποίησε στις 27 Μαρτίου στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο μετά από τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου η Κομισιόν είχε αντιτάξει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο την κατανομή των κονδυλίων για τα αντίστοιχα μέσα είχε λάβει υπόψη δηλαδή αυτές τι περικόπες τώρα. Η πρόταση βρίσκεται στο τραπέζι, αλλά είναι κατανοητό ότι οι επιλογέ αυτές είναι δύσκολε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποβάλουμε προτάσεις εντό των, των ανώτατων ορίων του MFF. Γι' αυτό το λόγο ε, βλέπουμε σημαντικές περικοπέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να τηρήσει τις τεράστιες ε, πολιτικές ισορροπίες στο βαθμό του δυνατού και τι πολιτικέ προτεραιότητε για το ΙΕΝΑ, για το DCI, για την ανθρωπιστική βοήθεια που αυξάνεται παρόλα αυτά σε σχέση με το 2013 παρά τη σημαντική μείωση του ανώτατου ορίου. Πρόκειται λοιπόν για μια δύσκολη άσκηση και όπως καταλαβαίνετε όλοι, όλοι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με αυτά τα ανώτατα όρια. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες αναμέσω, αναχρηματοδοτικό μέσο, δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω για το ΙΕΝΑ λεπτομερώς, αλλά είμαι βέβαιος ότι αν το χρειαστείτε η Κομισιόν μπορεί να σας στείλει μια ε, γραπτή απάντηση αργότερα για πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε όσον αφορά τον προπολογισμό 2014. Δυστυχώς οι συνθήκες, οι περιστάσεις είναι δύσκολες, αλλά όπως καταλαβαίνετε η Κομισιόν δεν μπορεί παρά να κάνει μια πρόταση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου. Κύριε Σιγητά, θέλετε να απαντήσετε. Κάποιε κάποιες ερωτήσεις έχουν παραμείνει από αυτές που διατύπωσε η κυρία Μάκη. Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι προτεραιότητες για την Αρκτική. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια ερμηνεία όλα αυτά της συμφωνίας για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Έτσι, διότι υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι στο πολιετές πλαίσιο προβλέπεται αύξηση για την πολιτική των εξωτερικών δράσεων για αυτό το κεφάλαιο 4. Δεν δικαιολογείται στο πρώτο έτος να έχουμε 12,5% περικοπή. Είναι πολιτική επιλογή που έλαβε η Επιτροπή αυτή όλα τα χρόνια τίθεται το ίδιο θέμα δημοσιονομική. Περικόπτουν σημαντικές προτεραιότητες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 50 εκατομμύρια για τους, ε, την Παλαιστινιακή Αρχή, για τους πρόσφυγες και σε άλλα σημαντικά κεφάλαια. Για την πολιτική γειτονία, που είναι μια πολιτική πολύ σημαντική για την Ευρωβουλή. Και η πολιτική απόφαση σε σχέση με το Συμβούλιο είναι να πρικοδοτηθούν οι δράσεις στο εξωτερικό επίπεδο με κονδύλια που θα είναι στο ύψο των περιστάσεων. Μια και είμαστε παγκόσμιοι ε, παίκτες στην παγκόσμια σκηνή και οι νέε προτεραιότητες για τις οποίες έκανε λόγο ο πρόεδρος της Λιθουανίας, ε, ε, υπουργό Εξωτερικών για την Λιθουανική Προεδρία και στην πολιτική γειτονία μας πιέζουν διαρκώς και με ιδιαίτερο τρόπο. Είναι αποφασιστική σημασία σε αυτές οι πολιτικές για τη σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και δεν μπορούν να απαντηθούν αυτές οι προτεραιότητες και ανάγκες με περικοπές τόσο σημαντικέ στα κονδύλια αυτά. Πολιτική γειτονία μείον 14,5% μέσω σταθερότητας μείον 3,5% κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας 20% περικοπή. Πρόεδρε, τούτον λεχθέντων το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά του και τις ευθύνες του ως σκέλος αρμόδιο για τα δημοσιονομικά, αρμόδιο μαζί με το Συμβούλιο. Έχουμε αυτό το δικαίωμα και το λογικό, αυτό που απαιτούν οι πολίτες μας είναι αυτό, να υπάρξει ένα περιθώριο ερμηνείας στο οποίο συνεισφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αποφασιστικό τρόπο όπως το κάναμε την προηγούμενη προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Θα προτείνω στα μέλη μια τακτική, ένα τακτικό ελιγμό να αποκαταστήσουμε αυτά τα κονδύλια στο προσχέδιο της Επιτροπής. Ένα πράγμα είναι ο εξορθολογισμός ε, στο επίπεδο των δεσμεύσεων και άλλο πράγμα είναι μια σε βάθος σημαντική περικοπή που δεν μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας στον τομέα των εξωτερικών δράσεων και στη συνέχεια περιπλέκεται η κατάσταση γιατί προστίθεται ένα επιπλέον στοιχείο για εφέτος. Υπήρξε αλλαγή στην ονοματολογία σε σχέση για παράδειγμα με την ε, ε, πολιτική που ακολουθούμε για τα αντικείμενα τα οποία παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αποτελέσματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν με την αλλαγή ονοματολογίας να δούμε με σαφήνεια τι γίνεται με τις περικοπές ε, στα κονδύλια για τις πολιτικές μας αυτές. Γι' αυτό σε σχέση με τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης για την πολιτική γειτονία και κυρία Γιάτεν Μάκη υπάρχουν εδώ λάθη διότι αυξήθηκαν τα μέσα, εδώ έχουμε το μέσο προένταξη που ε, λαμβάνει περισσότερες χώρες και με μικρότερο ποσό κιόλας. Γι' αυτό σας δίνω το παράδειγμα αυτό έχουμε ένα πολύ πιεστικό περιοριστικό χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά αυτά τα ποσά. Δυστυχώς θα πρέπει να τοποθετηθούμε με το ρυθμό που απαιτεί η Επιτροπή Προϋπολογισμού προτού το Συμβούλιο Υπουργών ε, τελεσίδικα τοποθετηθεί. Και γι' αυτό λοιπόν το Σεπτέμβριο θα πρέπει να εξεταστούν όλα αυτά τελεσίδικα. Θέλω να πω στην κυρία Γκόμες ότι συμμερίζομαι πολλές από τι ανησυχίε που εξέθεσε. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση ώστε να είναι ικανοποιητική για αυτές τις ανησυχίες που εξέφρασε, που τις μερίζομαι κι εγώ και είναι νόμιμες και θεμητές. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε πριν από τις ε, διακοπές ε, για το καλοκαίρι, τις θερινές διακοπές, οι σκιώδεις εισηγητές, μία θέση για να ψηφίσουμε μία, ένα τακτικό ελιγμό ως Επιτροπή για να δούμε τι θα πρέπει να γίνει μέσα στο πλαίσιο αυτών των περιορισμών και προσαρμογών να καθορίσουμε προτεραιότητες, μπορούν να γίνουν θυσίες, αλλά πρέπει να βρούμε και τη γραμμή με την οποία θα πορευτούμε. Αν αρχίσουμε να δεχόμαστε τέτοιους περιορισμούς δεν θα φτάσουν τα κονδύλια στο τέλος. Θα είναι ακόμα περισσο... λιγότερα αυτά τα κονδύλια από ό,τι οι ανάγκες μας. Αυτές είναι οι προθέσεις μου και οι προτάσεις μου Πρόεδρε. Και ευελπιστώ ότι μπορεί η Επιτροπή ενωμένη να προασπίσει τα συμφέροντα στην πολιτική εξωτερικών υποθέσεων. Διότι ένα στοιχείο επιπλέον έχουμε τη συζήτηση των διαφορετικών μέσων εδώ. Όχι μόνο την πολιτική στο εξωτερικό επίπεδο αλλά και τις πολιτικές σε άλλα κεφάλαια του προπολογισμού. Και βρίσκονται εδώ διαπραγματεύσεις ε, σε σχέση με συγκεκριμένες κοινέ κοινωνικές πολιτικές της Ένωσης που έχουν καθορισμένα ποσά, προκαθορισμένα ποσά. Δεν θα ήθελα οι προσαρμογές να γίνονται εις βάρος ε, της πολιτικής εξωτερικών υποθέσεων, όπου ε, έχουμε προβλήματα τα οποία τίθενται σαν συνέπεια άλλων ε, κινήσεων σε άλλα κεφάλαια. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Σημείωσα πολύ καλά τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι σκιώδεις εισηγητές της φιλελεύθερης ομάδας και η κυρία Γκόμες σκιώδης εισηγήτρια της σοσιαλιστικής ομάδας και ελπίζω ότι με τις τροπολογίες θα μπορέσουμε να βρεθούμε βρεθούμε στο ύψος των φιλοδοξιών μας ως Επιτροπή. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Και περάσουμε στο επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο θα ζητηθεί και κλεισμένο των θυρών. Να ζητήσω λοιπόν οποιονδήποτε δεν είναι ευρωβουλευτής ή μέλος του προσωπικού να εγκαταλείψει την αίθουσα. Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ.